ψηφίσματο τροπολογία 55 απορρίφθηκε «55 απορρίφθηκε». Η υπαριθμόν 43 απορρίφθηκε. 96. Επίσης απορρίπτωτα. Πενήντα επτά. Απορρίπτεται. Σαράντα τέσσερα. Απορρίπτεται. παριθμών 29. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 80. Απορρίπτεται. Υπαριθμών 58. Εγκρίνεται. 13. Απορρίπτεται. Σαράντα εννέα. Εγκρίνεται. Πενήντα εννέα. Απορρίπτεται. 60 απορρίπτεται. Δεκαπέντε απορρίπτεται. Δεκαεπτά πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 17. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Υπαριθμών 3. Απορρίπτεται. Τριάντα δύο. Απορρίπτεται. 61 Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα για την πρώτη δέσμη των τροπολογιών που αφορούν το κοινό ψήφισμα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την δεύτερη δέσμη τροπολογιών που αφορούν αυτή την κοινή πρόταση ψηφίσματος πρόκειται να ανακοινωθούν στις 8 και μισή. Στις 8 και μισή απόψε το βράδυ. Ακόμα γίνεται καταμέτρηση των ψήφων. Άρα στις 8.30 θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα για το δεύτερο τμήμα, για τη δεύτερη δέσμη τροπολογιών. Και τώρα αφού ανακοινώσαμε το αποτέλεσμα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την τρίτη ψηφορία. Έχουμε την ε, τρίτη δέσμη τροπολογιών όσον αφορά τη συντονισμένη δράση της Ένωσης για καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της. Όπως γνωρίζετε, η ψηφοφορία θα γίνει ακριβώς τον ίδιο τρόπο, όπως έγινε ε, και για την πρώτη και για την δεύτερη ε, φορά. Οπότε θα γίνει η ψηφοφορία μέχρι τις 6 ε, μετά μεσημβρία. Αρχίζουμε τώρα την ψηφοφορία και μέχρι τις 6 η ώρα, μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα θα διαρκέσει αυτή η ψηφοφορία. Τα δε αποτελέσματα για αυτή την τρίτη ψηφοφορία που γίνεται τώρα. Τα αποτελέσματα λέγω πρόκειται να ανακοινωθούν στις 10 και 50 το βράδυ. Άρα 8.30 τα αποτελέσματα και 10 και 50, 11 παρα 10 τα αποτελέσματα για την τρίτη ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας και διακοπή της συνεδριάσεως. Σας ευχαριστώ.